Då är Καλή σας. Καλό σας απόγευμα λοιπόν. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε. Έχουμε ψηφοφορίες, κάμουσες ψηφοφορίες. Και η πρώτη είναι ε, η ψηφοφορία για την επιχειρηματικότητα των γυναικών σε μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Η συγγήτρια είναι η κυρία Μαρίνα Γιανακουδάκη και η έκθεση ας ασχολείται με το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την αξία και το ρόλο της γυναικείας επιχειρηματικότητας όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη κτλ. Λοιπόν, η κυρία Γιανακουδάκη στην έκθεσή της αναφέρεται και σε κάποια εμπόδια τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες στον χώρο των επιχειρήσεων. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Γιανακουδάκη πριν να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επειδή πράγματι έχουμε πολλές ψηφοφορίες, θα προσπαθήσω να είμαι γρήγορη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με βοήθησαν στη σύνταξη της έκθεσης. Όλοι συνέβαλαν σημαντικά. Είναι σημαντική έκθεση για τις γυναίκες. Είναι μια ευκαιρία να ενισχύσουμε τις γυναίκες στο χώρο της επιχειρηματικότητας. Εκείνο που είναι σημαντικό επίσης ε, είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι η έκθεση είναι αρκετά έντονη. Δεν την αποδυναμώσαμε ασχολούμενοι και ασχολούμενες με άλλα δευτερεύοντα θέματα. Ελπίζουμε ε, λοιπόν να δείξετε και κάποια ανοχή θέλετε σε σχέση με κάποιες Μπας περιπτώσει να μην υπερψηφίσετε ε, τροπολογίες οι οποίες έχουν σαν στόχο να αποδυναμώσουν την έκθεση. τρία, σε τρία πράγματα αναγκάστηκα να πω όχι ήδη. Ε, το ένα θέμα είναι οι γυναίκες Ρωμά που δεν σημαίνει ότι δεν είναι σοβαρό το το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό αλλά θεωρούσα ότι θεώρησα ότι δεν ότι θα άλλαζε το χαρακτήρα της έκθεσης αν προσθεθόταν εδώ Η, μετά έχουμε τροπολογία 119 η ε, τροπολογία της Προέδρου ζητώ συγγνώμη αλλά δεν ε, μιλάμε ε, και αναφέρεται η τροπολογία αυτή στις α, ποσοστώσεις γυναικών, δεσμευτικές ποσοστώσεις γυναικών και ανδρών στα διοικητικά συμβούλια εταιριών κτλ. Κοιτάξτε να δείτε, δεν λέω ότι δεν έχετε δίκιο. Όμως εδώ μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν μεγάλα διοικητικά συμβούλια και όπου πραγματικά δεν μπορούμε να αναφερόμαστε σε αυτού του είδους τι ποσοστώσεις. Γι' αυτό δεν μπορώ να αντιδεχθώ. Επίσης η τροπολογία 165 που αναφέρεται στους στόχους που πρέπει να έχουμε για τη συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια. 169 επίσης, αριθμητικοί στόχοι. Δεν το δέχομαι ούτε αυτό. Ας παραμείνουμε σε αυτά που λέμε στην έκθεση για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ και τον προτέρων για την υποστήριξή σας. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γιάννα Κουδάκη. Η κυρία Κράτσα ζήτησε Ευχαριστώ πολύ Ε, ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γιανακουδάκη για όλη την εργασία που έκανε και για την ανταλλαγή απόψεων που ήδη και ακόμη και τώρα τελευταία στιγμή έχουμε. Ε, για την τροπολογία 165 ήθελα να πω. Επειδή εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Από τη μια μεριά είναι το πολιτικό μήνυμα, αν θέλουμε, σε αυτά τα, τα σώματα, τα bodies που είναι ε, τε, τα, της κατεύθυνσης της ε, αν πρέπει να υπάρχει ισορροπημένη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών. Επειδή ενοχλεί το... έχει μεταφραστεί στα γαλλικά και σε άλλες γλώσσες σαν διοικητικά συμβούλια και επειδή οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν αυτό τη μορφή, πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσουμε, και ίσως η γραμματεία μπορεί να επιμεληθεί στις μεταφράσεις, ε, να κρατήσουμε το Management Boards που είναι στα αγγλικά, ό,τι και αν σημαίνει όποιο είναι το όργανο διοίκησης και διεύθυνσης μιας επιχείρησης, έστω μικρής. Και οι μικρές επιχειρήσεις έχουν ένα όργανο κατεύθυνσης. Η ευχή λοιπόν της τροπολογίας είναι για ισόρροπη συμμετοχή χωρίς να, να βάζει συγκεκριμένο ποσοστό και στόχο. Απλά ήθελα να κάνω αυτή τη διευκρίνηση, διότι είναι κρίμα να παγιδεύονται κάποιοι συνάδελφοι ε, στο πώς χαρακτηρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο και αν είναι έτσι στις μικρές, στις μεσές και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κράτσα. Και ας αρχίσουμε τώρα την ψηφοφορία. Συμβιβασμός 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, Συμβαστική λύση 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 Α, θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για τροπολογία 57 Παρακαλώ ψηφίστε 57 EPP has one more. Το ΕΛΚ έχει μία επιπλέον ψήφο. The vote is Πέρας της ψηφοφορίας και απορρίπτεται 16 κατά 14 υπέρ. Πάμε στην τροπολογία 59 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται συμβαστική λύση 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική λύση 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε την τροπολογία 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 συμβαστική λύση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και συμβαστική λίστα 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική λίστα 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, 17, συμβαστική τροπολογία 17, εγκρίνεται, τροπολογία 88, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, συμβαστική τροπολογία 18, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 19, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, τροπολογία 96, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και προχωρούμε με την τροπολογία 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 Ωραία. Για την 118 λοιπόν ηλεκτρονική ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίνεται η 118, 16 υπέρ, 12 κατά. Προχωρούμε στην 119 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μπορούμε να το ελέγξουμε το αποτέλεσμα. 165 παρακαλώ. The vote is Πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίνεται 22 υπέρ 11 κατά. Προχωρούμε λοιπόν στη συμβαστική τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 124 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι πρέπει να το επαληθεύσουμε αυτό. 124 λοιπόν ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας Ισοπαλία 16 υπέρ 16 κατά απορρίπτεται. Α! You vote in favor. Yes. So... Α, εσείς ψηφίζετε υπέρ. Πολύ ωραία, Εγκρίνετε τότε. Now we go on amendments 125. Προχωρούμε στην 125 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ωραία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 125. Και όντω απορρίπτεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ωραία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 126. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τοπολογία 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 133 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 140 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ωραία, ωραία. Ελεκτρονικά για την 142. The vote is closed. Εγκρίνεται λοιπόν βάσει των αποτελεσμάτων. Τώρα πάμε στην συμβαστική τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 ε, καταπίπτει 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ωραία ελέγχουμε την 162 ψηφίστε closed Εγκρίνεται. 163 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 164 καταπίπτει 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 167 καταπίπτει 168 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ωραία Ελεκτρονική ψηφοφορία για την 169. Vote is closed. ψηφοφορίες και εγκρίνεται τελικά. 169. Τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Όχι. Do you want to vote on block? Amendments 1 and 2, Amendments 5. Να τις ε, ψηφίσουμε από κοινού 1 έως 5. 1 έως 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Πολύ καλή πρόταση να τις ψηφίσουμε από κοινού. Τώρα συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές καλύτερα να το ελέγξουμε Λοιπόν, η συμβαστική τροπολογία 3, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία και όντω συγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε την πέμπτη συμβαστική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 36 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ωραία, το ελέγξουμε. Την τροπολογία 36, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίες και εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 όχι. α, 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τροπολογία περιθμών 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα την τελική ψήφο παρακαλώ vote is closed and it's... Πέρας της τροπολογίας 29 ψήφι υπέρ, συγχαριστήρια κυρία Γιανακιού Κουδάκη. Thank you. And it's Mrs. Katza. Yeah. yeah. Ja, då gratulerar vi återigen Μάλιστα. Προχωρούμε. Συγχαρητήρια και πάλι κυρία Γιανακουδάκη. Και ερχόμαστε στην επόμενη ψηφοφορία τώρα. Οι γυναίκες και η δίκηση επιχειρήσεων είναι το θέμα της έκθεσης. Η συγγήτρια η κυρία Ρόδη Κράτσα. Η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική και συζητήθηκε πάρα πολύ, ήταν επίμαχη. Το θέμα είναι πώς μπορεί να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών στις επιχειρήσεις και συναντηθήκαμε και με ε, αρμοδίους το Μάρτιο για να ε, μάθουμε τι πρόοδοι έχουν επιτευχθεί ε, στο νομοθετικό επίπεδο. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Κράτσα για να κάνει κάποια σχόλια πριν περάσουμε στην ψηφοφορία. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε. Ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις συναδέλφους και τους συναδέλφους οι οποίοι με τις τροπολογίες τους, τις ιδέες τους, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έδειξαν για την έκθεση αυτή, ε, την εμπλούτησαν, έκαναν σαφή τη βούληση να στείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα καθαρό και ηχηρό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι είναι στιγμή πράγματι να ανοίξει συζήτηση και να πάρουμε δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν κράτη που έχουν ήδη προχωρήσει, έχουν πάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες που είναι ήδη σε εφαρμογή, αλλά κράτη είναι στο στάδιο τελικής επεξεργασίας. Υπάρχουν άλλα κράτη στα οποία έχει αρχίσει σχετική συζήτηση Υπάρχουν όμως και χώρες που δεν υπάρχει καμία δυναμική, κανένα διάλογος. Πιστεύω λοιπόν ότι το μήνυμα που θα στείλουμε εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεδομένης και της ε, δέσμευσης ε, για πρωτοβουλίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, θα δώσουν την ευκαιρία για μια ομοιόμορφη αντιμετώπιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και αν σεβόμαστε τις ιδιαιτερότητες, τις νομικές, τις πολιτισμικές, ε, των δομών των επιχειρήσεων που υπάρχουν στις διάφορες χώρες, αλλά μια ομοιόμορφη στρατηγική υπέρ της ενίσχυσης των γυναικών στα κέντρα που λαμβάνονται οι αποφάσεις οικονομικές στην αγορά, διότι η εμπειρία μας λέει σήμερα ότι δεν είναι μόνο θέμα αξιών και ηθικής, είναι ένα θέμα ε, επιδόσεων των επιχειρήσεων, είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να προσφέρει σε μια ανταγωνιστική κοινωνία και οικονομία που τόσο αναζητεί η Ευρώπη σήμερα. Ε, με τις συμβαστικές τροπολογίες ε, ε, προσπαθήσαμε να αντάξουμε τα πιο σημαντικά πράγματα ε, όπου στον κατάλογο ψηφοφορίας έχω βάλει αρνητικό πρόσημο είναι διότι υπάρχουν επαναλήψεις, είναι θέματα που δεν άπτονται ακριβώς του, του θέματος και του αντικειμένου. Ε, ευχαριστώ τις συναδέλφους όμως για όλη τους την προσφορά και τη συμμετοχή και ελπίζω θα έχουμε το αποτέλεσμα της πληροφορίας θα είναι ε, σαφές, ε, ηχηρό και αξιοποιήσιμο από την κοινωνία και από την πολιτική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Κράτσα. Η κυρία Κώστα ζήτησε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Πραγματικά επέδειξε μεγάλο πνεύμα συνεργασίας και ε, με μεγάλη προθυμία συζήτησε όλες τις προτάσεις και όχι μόνο από τη δική μας ομάδα. Νομίζω ότι κάναμε καλή δουλειά και θα βοηθήσουμε, θα δώσουμε μια όθηση τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και στα Εθνικά Κοινοβούλια στη συνέχεια και κύριο στην Ιταλία ψηφίζεται αυτό το καιρό ένα νομοσχέδιο προς την ίδια κατεύθυνση. Νομίζω λοιπόν ότι είναι όλο και περισσότερα τα κοινοβούλια που παίρνουν τέτοιες αποφάσεις και επίση πιστεύω ότι θα πρέπει να δείχνουμε πνεύμα επικοδομητικό και στις εκθέσεις πρωτοβουλίας. Δεν ζητάμε απλώ οδηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στη δίκη των επιχειρήσεων, αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια στους διορισμούς με βάση την αξιοκρατία, τα βιογραφικά και τα προσόντα των γυναικών αυτών. Επίσης, όχι μόνο στις ηγετικέ θέσεις, αλλά και στη βάση, σε χαμηλότερα απόσταση επιχειρήση. Είμαστε γενικά πολύ ικανοποιημένοι. Ευχαριστώ, κυρία Κώστα. Προχωρούμε στην ψηφοφορία. Ψήφι υπέρ της τροπολογίας 3, συμβαστικής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Με συμβαστική τροπολογία υπαρθών 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μισή τώρα. Η 40 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θα την ελέξουμε παρακαλώ τη 40 ηλεκτρονικά. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική υπαρήθευση. Πέρας. Όντως απερίφθη. Η συμβαστική 6 κατά αποχές εγκρίνεται. Η 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβιβαστική 5 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβιβαστική παρθόν 7 είπε. κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε τη τροπολογία παρθόν 59. Έτσι δεν είναι. Ε, Όχι. Συμβαστική Συμβιβαστική 10 πρώτα. Συμβιβαστική 10. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, τώρα. είναι η 59 η οποία καταπίπτει όμως. Και περνούμε στη συμβαστική αριθμών 8. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική υπαριθμόν 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 73 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 κατά πίπτη, 76 υπέρ. Τι, ποια θέλετε να ελέγξουμε, την 74. Αρχίζει η επαλήθευση για την τροπολογία 74. The vote is closed and it's adopted. Πέρας και εγκρίνεται. Λοιπόν, 76 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και πάλι έλεγχο θέλετε. 76. Αρχίζει η ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας, ορίστε, εγκρίθηκε. Η τροπολογία 53 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Θέλετε και εδώ έλεγχο. Αρχίζει για την 53. The vote is closed and it's adopted. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα η 86 νομίζω υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και η συμβιβαστική τώρα 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 100 εδώ έχει προφορική τροπολογία εισηγήτρια, την οποία βλέπετε στον κατάλογο ψηφοφορίας και μπορούμε να την ψηφίσουμε. Είπε, Κατά αποχές εγκρίνεται. 101 Είπε, Κατά αποχές απορρίπτεται. 102 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται η επόμενη καταπίπτει και θα περάσουμε στην 5 και την 6 μαζί. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα είναι η 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 13 υπέρ. Όχι 13. 13. Καταπίπτει η 13. Η 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 15 καταπίπτει. Η 16 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ Αντίθετα, η 17 έχει καταπέσει. Wait a moment, we must check. Μια πρέπει να ελέγξουμε κάτι. We could vote on amendment 17. Να ψηφίσουμε τη 17. Ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο για τη 17. Καλώ, αρχίζει η ψηφοφορία. 17. Η τροπολογία υπαριθμών 17. Πέρας. Απορρίπτεται, είπαμε. 18. υπε Κατά. Εποχέ. Εγκρίνεται. Τσεκ. Τσεκ. 18. Αρχίζει η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. 19. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21. Τσεκ. Για την 20. Ωραία. Ας την ελέγξουμε. Την 20. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 21. Υπέρ. Κατά αποχές. Α, όχι, καταπίπτει, λάθος έκανα. Άρα, 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 23 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 24 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τσεκ. Έφυγε 25. Καλώς. Αρχίζει η παλήθευση. Πέρας. Και απερίφθη. Και παίρνουμε στην 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ Α, έλεγχο. Yes. 28. So we vote on 28. 28 ψηφίζουμε. Συμφωνείτε να ψηφίσουμε την 28 υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. Number 10 with an oral amendment. Έχουμε την αιτιολογική αναφορά 10 με την προφορική τροπολογία ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία υπερθούν 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα έχουμε την τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. «25 υπέρ, Κατά αποχές κανένας κατά. Συγχαρητήρια κυρία Κράτσα. Μπράβο σας. Mrs. Jimenez wants the floor. Mrs. Jimenez wants the floor. κυρία Χιμένες θέλει το λόγο. it doesn't mean she changed her vote. No, it's 26 plus 7. Yeah, it's for voting. Yes, we have noted 26 voted in favor. Ναι, την υπερψηφίσαμε την 26. Όχι, 26. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πάντα ψηφοφορία γνωμοδότηση αυτή τη φορά για ε, το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην Επιτροπή Ελευθεριών που είναι αρμόδια καθήλυν. Ε, η κυρία Κώστα είναι η συντάκτριά μας για την γνωμοδότηση αυτή παρούσα και θα τη δώσω μέσα στο λόγο. Ναι. Θυμίζω μόνο και διευκρινίζω ότι μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας η επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτά τα θέματα αυξήθηκε. Και χάρη στη συνθήκη αυτή της Λισαβόνας έχουμε σήμερα την ευκαιρία να εγκρίνουμε μια τέτοια γνωμοδότηση που υποβάλλουμε στην Επιτροπή Ελευθεριών. Κατά πολέμηση, επαναλαμβάνω, του οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Κώστα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θίγονται οι γυναίκες από το οργανωμένο έγκλημα. Θα της δώσω λοιπόν το λόγο πριν περάσουμε στη ψηφοφορία. Ε, ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας Επιτροπής Ελευθεριών είναι μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες για το θέμα αυτό. Μετά τη συζήτησή μας για το δουλεμπόριο και τη διακίνηση ανθρώπων, ε, μιλούμε για ένα άλλο στοιχείο τώρα, μια άλλη πτυχή ε, του οργανωμένου εγκλήματος και της ε, καταπολέμησης του από τη δικαιοσύνη. Είναι πολύ φιλόδοξη αυτή η πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου, καλύπτει διάφορες πτυχές. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που βοήθησαν να εμπλουτιστεί το κείμενο συμφωνούμε πολύ συνάδελφοι για την ανάγκη. Ήταν τιμή συνεισφορά τους. Και ιδιαίτερα από τη σκοπιά των γυναικών. Στο οργανωμένο έγκλημα οι γυναίκες είναι κυρίως τα θύματα των δραστηριοτήτων αυτών. Του οργανωμένου εγκλήματος ιδιαίτερα για ε, αδικήματα ε, εις βάρος προσώπων. Και δεν θα πρέπει να είμαστε ουδέτεροι όταν μιλάμε για το οργανωμένο έγκλημα. Ουδέτεροι ως προς το φύλλο εννοώ, γιατί οι γυναίκες πλήττονται πάρα πολύ. Επίσης, οι γυναίκες ε, αγωνίζονται πάρα πολύ για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων, για την ατιμορρησία, κατά της ατιμορρησίας αρκεί να σκεφτεί κανείς πόσες γυναίκες δικηγόροι, δικαστές ε, αγωνίζονται. Και αξίζει να τις υποστηρίξουμε όσο γίνεται περισσότερο. Θυμάστε την οδηγία ε, για τη διακίνηση ανθρώπων. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πλέον να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δραστηριότητά της. θα οριστεί ένα συντονιστή που θα πρέπει από την αρχή να φροντίσει να εφαρμόζεται σωστά η οδηγία. Μια άλλη κατηγορία γυναικών που είναι θύματα και τι αναφέρουμε στο κείμενο είναι τα θύματα που είναι μάρτυρες ή συνεργάτες της δικαιοσύνης. Ε, ευχαριστώ την κυρία Χιμένεθ που προσέθεσε αυτό το σημείο. Πρόκειται για γυναίκες που λόγω της οικογενειακής τους κατάστασης είναι σε μια ενδιάμεση θέση, ε, δεν είναι ούτε θύματα ούτε συνένοχοι, αλλά γνωρίζουν καταστάσεις και πράγματα. Σκεφτείτε τη μαφία ή την καμόρα. Οπότε υπάρχουν ε, συστήματα προστασίας των γυναικών που γνωρίζουν αυτές τις δραστηριότητες, που τις απεμπολούν, που τις εγκαταλείπουν και συνεργάζονται με τη δικαιοσύνη, ακόμα και αν είναι στην ίδια τους οικογένεια. Ζητάμε λοιπόν να υπάρξει ένα νομοθετικό πλαίσιο πιο εναρμονισμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξασφαλίζεται καλύτερη προστασία των ε, θυμάτων και των μαρτύρων. Και ζητούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα η κυρία Ρέντινγκ που έκανε την εξαγγελία αυτή πολύ γρήγορα να φέρει το συνολικό νομικό πλαίσιο για την προστασία των θυμάτων. εντός αυτού του πλαισίου δεχτήκαμε κάποιες τροπολογίες για να ενισχυθεί η ε, γνωμοδότηση τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προβλέπουν κυρώσεις πιο αυστηρές και πιο ομοιογενείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβανομένων εδώ και ποινικών κυρώσεων. Στις περιπτώσεις που οι γυναίκες πέφτουν θύματα αυτού του είδους οργανωμένου εγκλήματος. Θα πρέπει να καταπολεμούμε κάθε είδους διάκριση και το κάνουν αυτό οι γυναίκες που εργάζονται στον τομέα της δικαιοσύνης. Γιατί ε, και η βία προκύπτει από τις διακρίσεις. Ψηφίζουμε. Η τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 14 Ψηφίζουμε τη 14. Μπορούμε να ψηφίσουμε μπλοκ όλες τις τροπολογίες από τη 15 μέχρι την 23. Συγγνώμη. Κυρία Γιανακουδάκη. Εγώ είμαι εντάξει μέχρι και την 20. Όχι παρακάτω. 15 με 20. In... amendment 16 is withdrawn. Yes, amendment 16 is withdrawn, you see that. 16 έχει αποσυρθεί. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. So on amendments Και συνεχίζουμε 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 25. Όχι, δεν καταπίπτει καθόλου. Η 14 16, συγγνώμη. Ψηφίζουμε την 25. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μπλοκ, μπορούμε να τα ψηφίσουμε από την 28 28 είπε, κατά εποχές απορρίπτεται. Την απορρίψαμε την 28. Α, θέλετε έλεγχο. Ωραία, αρχίζει τώρα για την 28. Πέρας. Α, εγκρίνεται τελικά. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ όχι μπλοκ δεν γίνεται δεν επιτρέπεται συνεχίζουμε 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα η τελική ψηφοφορία αρχίζει ηλεκτρονικά. The vote is closed. And it's... Πέρας, εγκρίνεται 29 υπέρ, κανείς κατά δύο εποχές, συγχαρητήρια κυρία Κώστα μου. Και το Σεπτέμβριο θα ψηφίσει η Επιτροπή Ελευθεριών. Mm. Och nu Συνεχίζουμε. Τώρα θα περάσουμε στην ψηφοφορία μια άλλη γνωμοδότηση προ την Επιτροπή Απασχόληση για την κινητικότητα και ένταξη ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης από την Επιτροπή μας προς την Επιτροπή Απασχόλησης είναι η Αντιπρόεδρος Μωρέν Σαρτιέ. Και θα τις δώσω αμέσως το λόγο. Ορίστε κυρία μου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι συζητήσαμε το πρωί την έκθεση και στην Επιτροπή Απασχόλησης και η δική μας συμβολή, στην Επιτροπή Γυναικών δηλαδή, αναμένεται με μεγάλη αδειμονία, διότι το πρωί μερικοί ήθελαν να τονιστεί ιδιαίτερα η δική μας συμβολή γιατί ο κύριος συντάκτης, ο αρμόδιος όπως στην ουσία είναι ο κύριος Κώσα ο οποίος τόνισε ότι εγκρίνει σχεδόν το σύνολο των προτάσεών μας που συμπληρώνουν λέει με πολύ χρήσιμο και συνεπή τρόπο τη δουλειά της Κοινωνικής Επιτροπής. Και γι' αυτό ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες για τη συμβολή τους στην επιτυχία αυτή και νομίζω ότι μεταξύ της Επιτροπής μας και της Επιτροπής Απασχόλησης θα έχουμε μια πολύ επικοδομητική και αποτελεσματική ελπίζω συνεργασία. Ωραία τότε. Θα συνεχίσουμε την ψηφοφορία. Υπάρχουν πολλέ συμβιβαστικέ προτάσει. Λοιπόν, η συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 έχει αποσυρθεί. Πάμε στην 6 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα η τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. το δεύτερο τμήμα τώρα της τροπολογίας 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13. Σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Α,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 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται είπα δεύτερο να απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, Όχι. εγκρίνεται. 45 υπέρ, α, θες, εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, θες, εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, θες, απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά, θες, εγκρίνεται. Ξανά έλεγχο στην 55, άρχεται η ψηφοφορία. Ξε... Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία το σύνολο, άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Συγχαρητήρια ομόφωνη έγκριση και 29 υπέρ. Σας ευχαριστούμε για όλη σας τη δουλειά. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Ιούνιο. Στο με... Τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο, Ιούλιο. Και στην Επιτροπή Απασχόλησης όμως τον Ιούνιο. Περνάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία γιατί είναι πολλές σήμερα, πολλές μας πέσανε. Λοιπόν, γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Απασχόλησης για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γνωμοδότηση αυτή μιλάει για θέματα ισότητος που αφορούν το όλο θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. και θέτει ορισμένα θέματα που εμποδίζουν, που την ελεύθερη κυκλοφορία των γυναικών. Λοιπόν, η κυρία Τσεσκόβα είναι η συντάκτρια, δυστυχώς όμως απουσιάζει. Γι' αυτό η κυρία Γιανακουδάκη θα μας πει δυο λόγια πριν αρχίσουμε την ψηφοφορία. Ορίστε κυρία Γιανακουδάκη μου. Ευχαριστώ. Θα διαβάσω απλώς αυτά που έγραψε η Αντρέα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης που συνεισέφεραν στη γνωμοδότησή μου και χαιρετίζω ιδιαίτερα την ευκαιρία να συζητήσουμε εδώ αυτό το σημαντικό θέμα. Το θέμα της κινητικότητας και ελεύθερης κυκλοφορίας είναι πολύ σημαντικό για ολόκληρη την Ένωση και από τα βασικά και θεμελιώδη δικαιώματα για τους πολίτες της Ένωσης να μπορούν να μετακινούνται από μία χώρα στην άλλη για να εργαστούν ή και για άλλου προσωπικού λόγου. Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν περισσότερες προσπάθειες για να μειώσουν το χάσμα μεταξύ των μισθών για τα δύο γέννη φύλλα και να μην υπάρχει παρεμπόδιση εργασίας από πολίτες μιας χώρας σε άλλη χώρα. Πρέπει οι εθελοντικές και δημόσιες υπηρεσίες να διευκολύνουν αυτή την κινητικότητα για τους ανθρώπους που εγκαθίστανται σε νέα χώρα να διευκολύνεται η πρόσβαση στην παιδεία των παιδιών τους και στις υγειονομικές υπηρεσίες. Ελπίζω η γνωμοδότησή μου να συμβάλλει σε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γανακουδάκη. Η κυρία Ζαμπόσκα έχει ζητήσει το λόγο. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Αν γίνεται θέλω να αποσύρω την τροπολογία μου 2 Υπάρχει όμως μία, υπάρχουν προφορικές τροπολογίες τώρα. Πρώτα οι τρία. Μπορούμε να ψηφίσουμε νομίζω και αυτές τις προφορικές τροποποιήσεις. Λοιπόν, τρία. Υπέρ. Against. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Number five. In Πέντε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έξι. Υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά και εγκρίνεται. 8 υπέρ. Α, έλεγχο έλεγχο του, της 7. Της 7. Επαλήθευση, άρχεται ψηφοφορία. Έληξε. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Ο επαλήθευση της 8. Άρχεται η ψηφοφορία. <clears throat> Έληξε. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. 12 υπέρ κατά εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση της 13 άρχεται η ψηφοφορία Ναι, έληξε, απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται επαλήθευση για την 16, 16. Επαλήθευση για 16 είπα κατά λάθος 17 αλλά εννοώ 16 άρχεται η ψηφοφορία τε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 έληξε, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα της 24 τώρα, η 25 υπέρ, κατά, αυτές εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, Ψηφίζουμε την 26 από την αρχή. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 όχι. Το δύο έχει αποσυρθεί. Έχει αποσυρθεί. Έχει αποσυρθεί. Α, ναι, έχει αποσυρθεί. Η κυρία Ζαμπόσκα το είχε πει. Η τελική ψηφοφορία λοιπόν του συνόλου. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικός. Ηλεκτρονικός πώς. Έληξε πανηγυρική έγκριση. Είπαμε. Στην Επιτροπή Απασχόληση τον Ιούνιο, στην Ολομέλεια τον Ιούλιο. σήμερα συνάδελφοι και συναδελφέ έχουμε ακόμα μία ψηφοφορία. Ακόμα μία και μετά. Μετά νομίζω ότι θα, ε, θα τελειώσουν. Λοιπόν, τελευταία και καλύτερη ψηφοφορία σχέδιο γνωμοδότησης για την εντολή για τριμερή διάλογο σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού 2012. Συντάκτρια ή συνεισηγήτρια είναι η κυρία Βαρβάρα Ματέρα θα υποβληθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών η γνωμοδότηση. Και μιλάει, κάνει λόγο για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να κινητοποιήσουμε περισσότερους πόρους για να μπορεί η Κομισιόν να εφαρμόσει την ποιοτική της πολιτική για την ανέχεια των γυναικών, για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε το πρόγραμμα Δάφνη, το Ίδρυμα των Φίλων κτλ. Έχει αμέσως το λόγο η κυρία Ματέρα που μπορεί να θέλει να πει δυο λόγια πριν αρχίσει η τελική ψηφοφορία μας. Κυρία Ματέρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Λυπούμε που ήρθα με κάποια καθυστέρηση γιατί είχαν λυμμένη υποχρέωση σε άλλες επιτροπές και αναγκάστηκα να έρθω τρέχοντας ασθμένουσα. Η γνωμοδότηση αυτή προς την Επιτροπή προπολογισμών είναι σημαντική διότι πρέπει να τονιστεί η πληροφόρηση που πρέπει να στέλνεται στα κράτη-μέλη κάθε χρόνο τακτικά. Προγράμματα σαν το Δάφνη είναι από τους κύριους στόχους της Επιτροπής μας για να καταπολεμηθεί η οικιακή βία κατά των γυναικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την Αντιπρόεδρό μας. Η κυρία Ζαμπόσκα έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λυπούμε που ξέχασα προηγουμένως να πω ότι και σε αυτή τη γνωμοδότηση θέλω να αποσύρω τις τροπολογίες μου 10, 18 και 19. 10, 18 και 19. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ζαμπόρσκα. Αρχίζουμε λοιπόν. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται 6 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται 7 υπέρ κατά εποχέ. εγκρίνεται 8 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται όχι επαλήθευση του 8 επαλήθευση της 8 άρχεται η ψηφοφορία για την 8 έληξε, εγκρίνεται τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 10 έχει αποσυρθεί από την κυρία Ζαμπόρσκα, η 11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 έχει αποσυρθεί και αυτή. Πώς επαλήθευση της 11 μάλιστα. Επαλήθευση της 11 άρχεται η ψηφοφορία. 11 έληξε η ψηφοφορία. Έχει αποσυρθεί. Έχει απο... απορριφθεί. Τώρα τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ σε δύο τμήματα, σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα 20 Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. ΧΕΣ εγκρίνεται. Θα ελέγξουμε την 21. Επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία. Για την 21 έληξε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται 23 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται χωριστά για την παράγραφο 11 ψηφίζουμε το σύνολό της χωρίς την έκφραση for EU funded measures υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα αυτή την έκφραση for EU funded measures υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, και εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, τα, χες, εγκρίνεται. Επαλήθευσης του δευτέρου τμήματος της 26 άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε, εγκρίνεται. Η τροπολογία 27 υπέρ, κατά, ποχές, απορρίπτεται. Επαλήθευση, επαλήθευση της 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται και τώρα η τελική ψηφοφορία για το σύνολο ηλεκτρονικά έρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Ματέρα μου. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ όλους και όλες. Όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία που εργαστήκαμε τόσο αποτελεσματικά σε αυτές τις ψηφοφορίες. And now we have this, and we have the postponed number five, and after that, coordinators. Yes, the first single mothers. Συνάδελφοι, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το επόμενο θέμα τη ημερήσια διάταξης. Υπάρχουν ακόμη μερικά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε σήμερα. Λίγη ησυχία παρακαλώ. Okej. Då går vi till ärende 13 på föredragningslistan. Σημείο 13 της σημερινής διάταξης. για την κατάσταση των μητέρων που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους. Παρακαλώ, επειδή πρέπει να συνεχίσουμε, αν θέλετε να κουβεντιάσετε κάτι άλλο, βγείτε από την αίθουσα. Λοιπόν, κατάσταση των μητέρων που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους η συγγήτρια η κυρία η αντιπρόεδρος μας η κυρία Ματέρα έχετε κυρία Ματέρα το λόγο για να μας κάνετε μια εισαγωγή για το, την έκθεσή σας πρωτοβουλία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σα ζητήσω πρώτα πρώτα να κάνετε λίγο υπομονή. Πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα. Για πρώτη φορά ασχολείται το Κοινοβούλιο με το ζήτημα αυτό και πραγματικά ε, τους τελευ τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες ε, δούλεψα σκληρά για να συντάξω την έκθεση αυτή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά ασχολείται με το θέμα. Δεν θα μπω σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά θα τονίσω μερικά σημεία τα οποία θεωρώ σημαντικά. Πρώτα-πρώτα, εδώ μιλάμε για τις μόνες μητέρες. Δεν μιλώ γενικότερα για τις μονογονικές οικογένειες. Ε, και ήρθα σε επαφή με μητέρες που μεγαλώνουν με μόνες τα παιδιά τους ήρθα σε επαφή με ε, συλλόγους ε, των μητέρων αυτών για να δω ακριβώς τα προβλήματα όχι μόνο βέβαια στη χώρα που βρισκόμαστε εδώ αλλά στη Γαλλία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Πολωνία ήρθα σε εποφή την περασμένη εβδομάδα κιόλας με νόσεις που όχι πλώς που των οποίων μέλη είναι μόνες μητέρες, αλλά που στηρίζουν και προσπαθούν να βοηθήσουν τις γυναίκες αυτές. Ε, Επίσης ήρθα σε επαφή με τους συλλόγους στήριξης ή και ε, μόνον μητέρων εδώ στο Βέλγιο με άλλα λόγια προσπάθησα να συλλέξω εμπειρίες, να συλλέξω απόψεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μόνες μητέρες για να μπορέσω να καλύψω τις διαφορετικές τις απόψεις που μπορεί να υπάρχουν και τις, ε, ε, στην έκθεσή μου. Δυστυχώς πρέπει να πω ότι οι γυναίκες οι οποίες μόνες μεγαλώνουν τα παιδιά τους, ε, ο αριθμός των γυναικών αυτών αυξάνεται στην Ευρώπη. Ε, στην ε, Βαρσοβία και στην Ιταλία που, όπου και τις αναφέρω αυτές γιατί είναι καθολικές χώρες όπου ενδεχομένως οι η θέση των γυναικών αυτών είναι κάπως διαφορετική ε, ο αριθμός αυξάνεται ταχύτατα η θέση τώρα των πολιτικών στη Βόρεια Ευρώπη, στη Δανία, στην, ε, και στη Γαλλία, μέχρι τη Γαλλία, όταν λέω Βόρεια Ευρώπη, ε, εδώ και χρόνια προσπαθούν και να βοηθήσουν και ασχολούνται με το ζήτημα αυτό και έτσι έχουν δημιουργηθεί δίκτυα α, στήριξης των γυναικών αυτών. Στη Νότια Ευρώπη, στη Μεσογειακή Ευρώπη, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα ε, Τέτοια δίκτυα δεν υπάρχουν. Η διαυρημένη διευρυμένη οικογένεια ε, είναι αυτή η οποία ε, αναλαμβάνει αν θέλετε την προστασία και τη στήριξη της μόνης μητέρας. Ε, α, πολλές γυναίκες που πρέπει να μεγαλώσουν μόλες τους τα, τους, τους, τα παιδιά τους γυρνούν στο πατρικό τους, στην οικογένεια τους αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στην Νότια Ευρώπη δεν θα χρειαζόταν ε, περαιτέρω θεσμική στήριξη αν θέλετε. Βεβαίως και στο βορρά και στο νότο και οπουδήποτε και να υπάρχουν οι γυναίκες αυτές είναι ευάλωτες η κατάστασή τους βεβαίως είναι μια προσωρινή είναι προσωρινή κατάσταση, διότι μπορεί στο μέλλον οι μητέρε αυτές να μην είναι μόνες τους, να βρουν κάποιο σύντροφο. Πάντως φαίνεται ότι για ορισμένους το προσωρινό της κατάστασης της μόνης μητέρας ε, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αφιερωθούν πόροι α, οικονομικοί ή άλλοι για τις γυναίκες αυτές. Υπάρχουν και χώρες όπου οι μόνες μητέρες στιγματίζονται και κατηγορού επικρίνονται ως ανεύθυνες νέες γυναίκες ε, ενώ και αυτό σίγουρα δεν είναι σωστό. Πρώτα πρώτα δεν είναι μόνο νέες γυναίκες. Υπάρχουν πάρα πολλές μόνες μητέρες ε, πάνω από την ηλικία των 25 χρονών και μέχρι τα 60. Ε, επίσης ε, δεν ε, είναι δεν θα νομίζω ότι η κατηγορία της ανευθυνότητας επίσης δεν ισχύει Ωστόσο στιγματίζονται από την κοινωνία όπως έλεγα και με μια έννοια τιμωρούνται κιόλας. Από εκεί και πέρα οι μόνες μητέρες δεν είναι σίγουρο ότι έχουν πάντα ένα μόνο παιδί, ίσως αυτή είναι η καλύτερη περίπτωση. Υπάρχουν όμως και μητέρες που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους και έχουν πάνω από ένα παιδί. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα και όχι μόνο σχετικά με την αδυναμία να δουλέψουν οι γυναίκες αυτές αλλά και προβλήματα μεταξύ των παιδιών η, η δυσκολία πάντως της πρόσβασης σε θέσεις εργασίας ε, είναι πραγματικά σοβαρό ε, πολύ δύσκολη ή πολύ σοβαρή. Συγγνώμη. Όσον αφορά τώρα την υγεία των γυναικών αυτών, βλέπουμε ο, στατιστικά τουλάχιστον ότι οι γυναίκες αυτές ε, επειδή πιέζονται ίσως περισσότερο στην καθημερινή του ζωή επειδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες υγείας ε, βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση υγείας από τις άλλες γυναίκες αντίστοιχη ηλικία. Το άλλο χαρακτηριστικό της κατηγορίας αυτής της ε, γυναικών είναι ότι οι μη καλά μορφωμένες γυναίκες ε, είναι περισσότερες στην κατηγορία αυτή και γι' αυτό αντιμετωπίζουν και δυσκολίες ακόμη μεγαλύτερες από τις υπόλοιπε γυναίκες ε, στο να βρουν δουλειά. Οι περισσότερες και λόγω της ε, ανάγκης να φροντίσουν για τα παιδιά αλλά και λόγω του μορφωτικού τους επίπεδου αναγκάζονται να περιορίζονται σε μερική απασχόληση. Στο δεύτερο μέρος της έκθεσής μου Αναφέρομαι τώρα όχι στην περιγραφή, αναφέρομαι όχι στην περιγραφή μοναχά των ε, γυναικών αυτών, αλλά και στο τι θα μπορούσε να γίνει για τις γυναίκες αυτές. Ενθαρρύν, λέμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, φροντίσουν να προστατεύσουν τις γυναίκες αυτές να τις φέρουν σε επαφή σε, με οργανισμούς, ενώσεις, συλλόγους που θα μπορούσαν να τους στηρίξουν και ενδεχομένως να ήταν καλό να συνεργαστούν και μεταξύ τους τα κράτη-μέλη για να βοηθήσουν ακόμη καλύτερα. Ίσως αυτό είναι πιο σημαντικό στην Νότια Ευρώπη. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε πολιτικές σε εθνικό επίπεδο που παρέχουν έμεση βοήθεια, αν θέλετε. τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν μέσα στα πλαίσια της καταποτε... καταπολέμησης της φτώχειας να εντάξουν και τις γυναίκες αυτές και να εφαρμόσουν αντίστοιχα μέτρα τα οποία δεν είναι άμεσα επιδόματα αλλά είναι βοήθεια για πρόσβαση σε κάποια βασικά τρόφιμα παραδείγματο χάρη. Από την άλλη μεριά υπάρχει η... ίσως θα πρέπει να θεσπιστούν και ε, φορολογικά μέτρα και φορολογικές διευκολύνσεις για τις γυναίκες αυτές, σαν και αυτές που προβλέπονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ολλανδία. Ή επίσης θα μπορούσαν, θα μπορούσαν να αναζητηθούν ε, φάνταστες λύσεις για να αναπληρωθεί τρόπον την η έλλειψη του δεύτερου γονέα θα μπορούσε στο, για το θέμα αυτό να γίνει κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι, οι μόνες μητέρες δεν είναι απλά μόνες φτωχές γυναίκες γιατί αυτή η σύγχυση πολύ συχνά γίνεται οι μόνες μητέρες είναι γυναίκες οι οποίες έχουν παιδί ή παιδιά που συνήθως ζουν με δύο γονείς αυτά τα παιδιά αυτή τη στιγμή ζουν με ένα γονιό μονάχα και γι' αυτό ίσως θα έπρεπε να αναζητηθούν λύσεις όπως παραδείγματο χάρη να ενθαρρυνθούν επιχειρήσεις, εταιρείε να ε, προσλαμβάνουν μόνες μητέρες τις οποίες όμως θα στηρίζουν αν πρέπει να διακόψουν την εργασία τους ή θα, οι οποίες θα μπορούν να, να καλύπτουν αν θέλετε και τη φροντίδα του παιδιού μέσω των εταιριών αυτών στην Ολλανδία η οι μόνες μητέρες ε, δεν χρειάζεται να πληρώσουν για την ιατρική παρακολούθηση και περίθαψη των παιδιών τους. Έχουν, όπως είπαμε προηγουμένως, και φορολογικές διευκολύνσεις και προσπαθούν ε, επιλέγονται κατά προτίμηση σε θέσεις εργασία όπου μπορούν να δουλεύουν από το σπίτι Α, και αυτά τέτοιου είδους λύσεις, τέτοιου είδους μέτρα είναι θετικά κατά την άποψή μου και για τις γυναίκες. Αυτές και για τις επιχειρήσεις και τις οποίες δουλεύουν, αλλά και για την κοινωνία γενικότερα. Επίσης η δυνατότητα χαμηλότερων ενοικίων παραδείγματος χάρη ε, βοήθεια από το κράτος, επιδοτήσεις ενοικίων. Τέτοιου είδου ιδέες χρειάζονται και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο του πιστεύω ότι θα επικριθώ για πάρα πολλά από αυτά που προτείνω στο σχέδιο έκθεση που έχετε στη διάθεσή σας ε, Υπάρχουν όμως κάποιες χώρες τις οποίες τα πράγματα είναι καλύτερα για τις μόνες μητέρες, όπως τη Γερμανία παραδείγματος χάνει σε σχέση με εργασιακά θέματα ή ε, θέματα απασχόλησης σε μπαση περιπτώσει. Ε, και άλλες χώρες στις οποίες η κατάσταση είναι κακή. Και αυτό είναι λίγο άδικο. στις επαφές που έκανα προετοιμάζοντας την έκθεση αυτή ήρθα σε επαφή με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών ε, όχι από όλες τις χώρες βεβαίως που δεν είναι λόγο α, και ένα από τα παράπονα που φαίνεται να έχουν οι γυναίκες αυτές είναι ότι δεν υπάρχουν οργανισμοί, δεν υπάρχουν ομάδες πίεσης υπέρ αυτών. Και ζήτη, μου ζήτησαν αν είναι δυνατόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δράσει σαν ομάδα πίεση πίεσης υπέρ των γυναικών αυτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Ματέρα, λέει η Πρόεδρος και τώρα η κυρία Γιάρογκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Επιτέλους ε, ε, ερχόμαστε, αρχίζουμε να ασχολούμεθα με αυτό πιο συγκεκριμένα για τα τελευταία έξι χρόνια συζητιόταν στα παρασκήνια με μη κυβερνητικέ οργανώσεις κτλ. Χαίρομαι που συζητούμε λοιπόν το, το θέμα αυτό και Ξέρω βεβαίως τι ήδη έχουν γίνει και πράγματα υπέρ των μόνων μητέρων από κάποιες επιχειρήσεις. Θυμάμαι ε, το Marks and Spencers και ε, εκπροσώπους από την εταιρεία αυτή που ήρθαν εδώ και μας μίλησαν για το τι γίνεται με τις μόνες μητέρες στο Λονδίνο και για το, ε, κάποιες πρακτικές ας πούμε που εφάρμοζαν εκείνοι και θα μπορούσαν να αντιγραφούν. Τώρα, να πω κάτι τι πριν από μερικά χρόνια, όταν πήγαμε σε κέντρα στα οποία μπορούσαν να προσφεύγουν νέες μόνες μητέρες. Ε, όταν πηγαίναμε εκεί λοιπόν είδαμε ότι οι περισσότερες από αυτές τις νέες γυναίκες ήταν οι γυναίκες που είχαν ε, κακοποιηθεί, που ε, έφευγαν από το σπίτι τους λοιπά Τώρα λόγω της οικονομικής κρίσης ε, δυστυχώς ο αριθμός των γυναικών αυτών αυξήθηκε και οι, κατηγόροι, οι γυναίκες που προσφεύγουν είναι άλλο είδους. Ε, δυστυχώς επίσης σε πάρα πολλές χώρες όπως τη δικιά μου έχουν, έχει μειωθεί ο αριθμός αυτών των κέντρων στα οποία μπορούν να προσφύγουν ε, οι μόνες μητέρες οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Οφείλουμε να δεχθούμε να οφείλουμε να ομολογήσουμε. Εδώ λοιπόν πρέπει να προσέξουμε ε, τι γίνεται. Και κάτι τι άλλο που χαίρομαι που το βάζετε στην έκθεσή σας αλλά δεν το είχαμε συζητήσει μέχρι τώρα είναι τι γίνεται ακριβώς στη, στο χώρο της απασχόλησης. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κάποιες μητέρες οι οποίες δρέπονται ή θεωρούν ότι καλύτερο είναι να μην πούν καν ότι είναι μόνες μητέρες όταν ζητούν δουλειά. Είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να γίνουν λίγο παρα, να γίνει κάπως παραπάνω έρευνα σε σχέση με αυτές τις γυναίκες μέσα από τα πλαίσια ίσης μεταχείριση των φίλων ή ε, μη διακρίσεων σε εθνικό επίπεδο γιατί ένα πράγμα είναι να πει κανείς ότι ε, είναι μόνη, είμαι μόνη μητέρα και ε, θέλω να μείνω στο σπίτι μου και πρέπει να μείνω στο σπίτι μου και άλλο είναι να πάει κανείς να ψάχνει δουλειά και να ε, ντρέπεται ή να προσπαθεί να το κρύψει γιατί ξέρει ότι θα είναι η πρώτη που θα απολυθεί ή που θα χάσει δουλειά τη θα, παρα... τεθεί στο περιθώριο μόλις υπάρξουν προβλήματα. Είναι πολλά λοιπόν ε, τα, είπατε ότι στιγματίζει η κοινωνία τις γυναίκες αυτές. Αυτό είναι γεγονός και πολλές φορές τα ψυχολογικά προβλήματα είναι πολύ πιο σημαντικά και ε, οδυνηρά από πρακτικά και οικονομικά προβλήματα. Η κυρία Παρανόβια. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Ματέρα για την εξαιρετική έκθεσή της. Είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα Όντως οι μόνες ε, μητέρες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και απομόνωσης και από, σχεδόν αποκλεισμού από την κοινωνία οπότε πρέπει να τα δούμε συνολικά τα προβλήματα και να καταβάλουμε πάσα προσπάθεια και εμείς και τα κράτη-μέλη ξεχωριστά το καθένα για να βοηθηθούν οι γυναίκες αυτές. Πράγματι το κομμάτι που σχετίζεται με τη φροντίδα των παιδιών είναι σημαντικό ε, Επίσης η δυνατότητα εκπαίδευσης μετεκπαίδευσης των μόνων μητέρων γιατί όπως ελέγχθη το μορφωτικό τους επίπεδο ή το, ή το εκπαιδευτικό τους επίπεδο είναι μάλλον χαμηλό υπάρχουν όμως και άλλες ανάγκες των μόνων μητέρων διαφορετικές σε κάθε χώρα που ίσως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με μέτρα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των γυναικών αυτών. Πράγματι και στο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό τομέα κάτι θα μπορούσε να γίνει για να μπορέσουν και οι γυναίκες αυτές μετά να ενταχθούν απόλυτα ε, και πλήρως στην αγορά εργασίας. Ε, εδώ παίζουν ρόλο βέβαια και τα κίνητρα για τους εργοδότες, ε, επιχειρήσεις, εταιρείες που θα μπορούσαν να κατά προτεραιότητα να χρησιμοποιήσουν τις γυναίκες αυτές για κάποιες θέσεις που θα μπορούσαν να έχουν βρεφικούς, βρεφονιπιακούς σταθμούς για να τις βοηθήσουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κάνει κάποια δουλειά στο παρελθόν ιδιαίτερα σε σχέση με την αύξηση της κοινοτικότητα των μόνων μητέρων ε, αλλά νομίζω από εκεί και πέρα ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τα, το έργο αυτό στην Στου, στους στόχους της Βαρκελόνης αναφέρονται επίσης πολλά θέματα που πρέπει να προωθήσουμε και όπου δεν έχει επιτελεστεί ε, σημαντική πρόοδος θα πρέπει να συνεχίσουμε. Θα πρέπει να δούμε και το θέμα της ε, φτώχειας, ε, αν είναι πιο εύκολο οι γυναίκες αυτές να πέσουν ε, στο επίπεδο της στόχης ή κάτω από αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερα που αναφερθήκατε και στην ανάγκη να γίνουν πράγματα για να αναπληρωθεί τρόπον την άγια απουσία του ο δεύτερου γονέα. Ευχαριστώ κυρία Παρβανόβα. Η κυρία Στρέλα τώρα έχει το λόγο. Muito obrigada, Presidente. Eu também gostaria de começar por Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια, την κυρία Ματέρα, για την δουλειά που έκανε. Η έκθεσή της δεν αναφέρεται μονάχα σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά αναφέρεται και σε κάποια ζητήματα πολύ βασικά και θεμελιώδη για τις γυναίκες. Αναφε... Ακούστηκαν στατιστικά στοιχεία. Πίσω από τα στατιστικά στοιχεία κρύβονται προβλήματα ε, ολόκληρων οικογενειών. Α, ολόκληρων στρωμάτων της κοινωνίας μας θα έλεγα οι μόνες μητέρες ε, είναι γυναίκες οι οποίες βρίσκονται μόνες τους με ένα ή περισσότερα παιδιά μετά από κάποιο διαζύγιο ή γυναίκες οι οποίες εγκατέλειψαν την οικογενειακή αιστεία λόγω κακοποίησης και τέτοιου είδους προβλημάτων. Οι καταστάσεις των μόνων μητέρων είναι πολλές και διαφορετικές και εξα... βεβαίως η κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη είναι διαφορετική όπως είπατε. Είπατε είναι διαφορετική κατάσταση στο βορρά α, από ότι από αυτή που παντά κανείς στο Νότο. Στην Πορτογαλία, παρόλο που βρισκόμαστε στο Νότο, υπάρχουν ακόμη πιο διαφορετικές καταστάσεις και στο εσωτερικό της χώρας μας. Ε, οι κατηγορίες, οι γυναίκες αυτές για τις οποίες μιλάμε ε, προέρχονται από από όλα τα κοινωνικά στρώματα, ε, ακόμη και οικονομικά εύρωστα κοινωνικά στρώματα που βρίσκονται μόνες τους με τα παιδιά τους μετά από ένα διαζύγιο και όπου ο πατέρας παραδείγματος χάρη δεν α, ε, καταβάλει τη διατροφή την οποία επέβαλε το δικαστήριο πατεράδες Υπάρχουν πολλοί πατεράδες που δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και που γι' αυτό οι μητέρες ξαφνικά από μία οικονομικά καλή κατάσταση ε, βρίσκονται σε μία κατάσταση φτώχειας σχεδόν τα παιδιά αυτά που συνήθισαν που μεγάλωσαν μέχρι ενό σημείου σε ένα αλφα κλίμα ξαφνικά βρίσκονται σε... και έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα τελείως διαφορετικά. Ε, επίσης, το τομέα της απασχόλησης είναι δύσκολο για πολλές από τις γυναίκες αυτές να βρουν δουλειά και ακόμη και αν βρουν δουλειά είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδυάσουν επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε όλοι μας για να στηριχθούν οι γυναίκες αυτές οι γυναίκες αυτές άσχετα από την κατάστασή τους, άσχετα από το επίπεδο μόρφωσή τους, άσχετα, από το κοινωνικό στρώμα στο οποίο ανήκουν. Το να βοηθήσουμε τις γυναίκες αυτές θα βοηθήσει στο να διατηρηθεί ε, η κοινωνική συνοχή. Το να βοηθήσουμε τις γυναίκες αυτές σημαίνει ότι βοηθούμε και τα παιδιά τους. Καταπολεμούμε τη φτώχεια. Τα και βοηθάμε τα παιδιά που είναι φτωχά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την κοινωνία μας. Και κλείνοντας γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω άλλη μια φορά την κυρία Ματέρα και είμαι στη διάθεσή της για να συνεργαστώ και στο μέλλον. Ευχαριστώ κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Ματέρα για την έκθεσή της. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι οι ανήπατρες μητέρες, εκείνες που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους, αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες από ό,τι οι οικογένειες. Πάντως στην έκθεση κάτι μου λείπει. Υπονοεί η έκθεση ότι όλες οι μόνες του μητέρε δεν έχουν μόρφωση, έχουν τρομερές αδειξότητες στη ζωή τους για να επιβιώσουν. Ενώ το κλειδί εδώ είναι διαφορετικό. Και ακούστηκε προηγουμένω ότι από χώρα σε χώρα διαφέρει και η κατάσταση αλλά και η νομοθεσία. Να σας πω πώς έχει η κατάσταση στη χώρα μου, στη χώρα των Βάσκων. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός ε, των ανήπαντρων μητέρων αυξήθηκε ε, σε μεγάλο βαθμό, αλλά είναι τελώς ε, διαφορετικές από αυτό που λέει η έκθεση. Οι εργάζονται, αποφασίζουν μόνες τους αν θέλουν να έχουν άντρα ή όχι και αποφασίζουν επίσης μόνες τους αν θέλουν να έχουν παιδιά, βιολογικά ή υιοθετημένα. Και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν αναφέρεται αυτή η πραγματικότητα στην έκθεση Ξέρω ότι έχουμε γυναίκες με δυσκολίες, αλλά κάπως πρέπει να κάνουμε και μία διάκριση, γιατί πολλέ φορέ είναι και επιλογή του. Επίσης για την ισότητα, αναφέρουμε και ε, αλλού αυτά τα θέματα, ας πούμε, ο συνδυασμός, η συμφιλίωση του οικογενειακού και του επαγγελματικού βίου είναι κάτι που έχει να κάνει και με τις ε, μόνες τους μητέρες, τις ανήπαντρες, αλλά και εκείνες που έχουν ε, οικογένεια. Δηλαδή, κάποιες γυναίκες που έχουν ε, ε άντρα, το 70% το επομίζονται οι ίδιες οι γυναίκες ακόμα. Ακόμα και αν δεν είναι μόνες τους. Την ίδια δυσκολία έχουν. Δηλαδή, στην έκθεση ε, αναφέρονται κάποια γενικά θέματα που είναι θέματα ευρύτερα ε, που άπτονται της ισότητας των δύο φύλων και όχι αποκλειστικά των μητέρων αυτών. Σε ό,τι αναφορά σε ό,τι αφορά, συγγνώμη, ε, τη υπόθεση αυτού του γενικού επιδόματος. Δεν το έχουμε συμφωνήσει. Υπάρχει ένα γονικό επίδομα, αλλά δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, μπορεί να αφορά και τις μητέρες και τους πατέρ που παίρνουν γονική άδεια. Η κυρία Στρέλα επίσης αναφέρθηκε στην περίπτωση της Πορτογαλίας. Εγώ μπορώ να σας πω ότι γίνεται όχι μόνο στο βασίλειο της Ισπανίας αλλά και στην αυτόνομη περιφέρεια της χώρας των Βάσκων που οι ανήπατρες μητέρες έχουν τη δυνατότητα να πάρουν επιδόματα από την περιφερειακή κυβέρνηση ή από την τοπική αυτοδιοίκηση και μάλιστα και μόρια για να παίρνουν κοινωνική στέγη. Όλα αυτά καλό θα ήταν να τα βάλουμε και στην έκθεση. Για, για να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου, μιλάτε για ποσοστά, για ανήπατρες μητέρες. Ακριβώς όμως επειδή διαφέρει η νομοθεσία από χώρα σε χώρα, υπάρχουν χώρες που επιτρέπουν σε άνδρες ανήπαδρους να ε, υιοθετούν. Ή επίσης ε, υπάρχουν ομοφιλόφιλα ζευγάρια που χωρίζουν και έχουν παιδιά. Τι θα γίνει ε, και πού είναι τα ποσοστά αυτά. Ίσως καλό θα ήταν η Επιτροπή μας να ε, κάνει μια προσπάθεια για να ενσωματώσει και την αυτή πραγματικότητα. Γίνεται λόγο για το 5%. Και τι γίνεται, επειδή είναι λίγοι πρέπει να του αφήσουμε απ' έξω. Ναι. Και το τελευταίο που είπε η κυρία Στρέλα. Εμείς θα πρέπει να σκεφτούμε την ευημερία και ε, την ευτυχία των παιδιών. Mm. Οπότε τι μας νοιάζει αν είναι ανήπαντρη μητέρα ή ανήπαντρος πατέρας ή μόνος του πατέρας ή μόνη της η μητέρα. Όταν νομοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι καλά το παιδί. Ανεξάρτητα από το ποσοστό, ακόμα και είναι μεγαλύτερο το ποσοστό των γυναικών. Και μην ανησυχείτε, θα κάνω και τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπιλμπάο. Η κυρία Τόμψεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Θα μιλήσω εξ ονόματος της κυρίας Γκουρμάη που είναι σκιώδης συγγήτρια και σήμερα κολλείεται γιατί είναι στην Πολωνία. Και θα σας πω και μερικά δικά μου σχόλια παρόδο, διότι συμφωνώ για τις πρωτοβουλίες ως προς το ωράριο και τα ε, ευεργετήματα ή τα επιδόματα ε, των ε, μητέρων που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους. Ε, αυτά μου φαίνονται λίγο παλιωμοδίτικα, γιατί ίσως είμαι η μόνη εδώ ανήπαντρη μητέρα και ξέρετε οι αντίπαντρες μητέρες είναι ε, η πιο γερή κρίκη της αλυσίδας στην κοινωνία. Είναι μόνες τους, παίρνουν πολύ σκληρές αποφάσεις, φτιάχνουν, διαμορφώνουν τη ζωή τους μόνες τους και αν δεν είναι σκληρές από την αρχή γίνονται σκληρές στην πορεία. Και επίση δεν θα πρέπει να υποτιμούμε αυτό που είναι η εργασία που ονομάζουμε οικιακά. Οι παντρεμένες γυναίκες πολλές φορές έχουν περισσότερη δουλειά ε, από τις ανήπαντρες. Ε, αλλά οι παντρεμένες ε, που λέτε ότι έχουν δουλειά μπορεί καμιά φορά το βράδυ να κάθονται δίπλα στο σύζυγό του στον καναπέ και να βλέπουν τηλεόραση. Ενώ οι ανήπαντρε κάθονται στον υπολογιστή και κάνουν ε, ε, διαλληλογραφίε μαθήματα να πάρουν κανένα μάστερ. Αυτά από μια ανήπαντρη μητέρα. Και θα σας διαβάσω τώρα τι μου είπε η συνάδελφο Ζήτα Γκορμάη να διαβάσω. Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή έχω άλλες ανηλυμένες υποχρεώσεις, δεν μπορώ να είμαι στο δεύτερο τμήμα της σημερινής συνεδρίασης. Επιτρέψτε μου όμως να αναφέρω μερικά θέματα και ερωτήσεις σχετικά με την έκθεση της αγαπητής φίλης και συναδέλφου Ματέρα. Γίνεται λόγος για χαμηλότερη μόρφωση και χαμηλότερη αμοιβή των ε, ανήπατρων Θα πρέπει να μιλώσουμε και για υποαπασχόληση όταν αναγκάζονται να εργάζονται σε ε, χαμηλότερες θέσεις εργασίας. Το θέμα της συμφιλίωσης ε, του εργασιακού με τον οικογενειακό βίο είναι ξέχον για τις ανήπαντρες μητέρες ή τις μόνες μητέρες. Το ξέρουμε όλοι, το λέει και η έκθεση και θα πρέπει όμως να ε, το αναλύει περισσότερο. Επίσης είναι σημαντικό να μιλήσουμε και στο διατακτικό, όχι μόνο στην αιτιολογική ε, έκθεση για το ρόλο των επιχειρήσεων να προσλαμβάνουν ανήπαντρε μητέρε. και δεν θα πρέπει ε, να φοβηθούμε να το γράψουμε και στο διατακτικό. Ανησυχώ λιγάκι από το πρόβλημα της φοροαπαλλαγής για τις ανήπαντρες μητέρες. Η φοροαπαλλαγή, η μείωση του φόρου, ε, ελάφρυνση, έχει να κάνει με το εισόδημα ε, και δεν θα πρέπει να τις αποκλείουμε από τα επιδόματα. Είναι κοινωνικό το ε, πρόβλημα και θα πρέπει να λυθεί με κοινωνικό τρόπο και με κοινωνικά επιδόματα. Καμιά φορά έχω την αίσθηση ότι η αιτιολογική έκθεση της ε, έκθεσης είναι πιο χαρακτηριστική και πιο εύγλωτη από το διατακτικό. Και προτείνω να πάρετε κάποιες ιδέες από αυτές τις παραγράφους, ε, από τα εκτιμώντα και να το βάλετε στην έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Σας φιλώ. Ζήτα Γκουρμάη. Ευχαριστώ κυρία Τόμσεν. Η κυρία Λούλη, παρακαλώ. Μάλιστα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα εισαγωγικό σχόλιο. Βλέπω λίγο τη γαλλική μετάφραση και νομίζω ότι χρειάζεται να τη χτενίσουμε λίγο γιατί δεν καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τη διατύπωση στα γαλλικά. Δεν ξέρω να σας τα πω ίσως και μετά. Δεν τα πολύ καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Ε, ε, ε, Συμφωνώ και με αυτά που είπε η κυρία Μπιλμπάο. Γιατί σήμερα στις κοινωνίες μας έχουμε νέα φαινόμενα. Και πριν από 30 και 40 χρόνια εγώ ήξερα γυναίκες που δεν ήθελαν να παντρευτούν ήθελαν να κάνουν παιδί, ένα παιδί και δύο παιδιά, αλλά όχι άντρα. Και δεν υπήρχε πρόβλημα, γιατί ήταν επιλογή τους ελεύθερη. Και δεν πέφτανε στη φτώχεια επειδή κάνανε ένα παιδί. Όλες οι ανήπαντρες ή οι διαζευμένες μητέρες οι χείρες και τα λοιπά που ζουν μόνες τους δεν είναι και πανφτωχές και εξαθλειωμένες. Ε, και ευτυχώς που δεν είναι. Δεν θα πρέπει να γενικεύουμε λοιπόν. Επίσης πρέπει να σας πω ότι διατέλεσα 15 χρόνια δήμαρχος στην πόλη μου και 30 χρόνια ήμουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί να δείτε τι έχουν δει τα μάτια μου σε ό,τι αφορά την κατάσταση των γυναικών. Και εγώ διαρωτήθηκα, τι περνάει από το μυαλό μιας γυναίκας και τι αίσθηση ευθύνη έχει μια γυναίκα που γεννάει τρία και τέσσερα και πέντε παιδιά με διαφορετικούς πατεράδες κάθε φορά, χωρίς να νοιάζεται για την κατάσταση των παιδιών αυτών. Πρέπει να σας πω ότι στη χώρα μου, δυστυχώς, δεν είναι τόσο πλούσια στο παρελθόν, έχουμε χτίσει συστήματα κοινωνικά που ευνοούνται οι ανήπαντρες μητέρες. Αν θέλει κανείς να υποφεληθεί από τα κοινωνικά επιδόματα ένα κατώτατο εισόδημα, συμφέρει πιο πολύ να τα παίρνεις αυτά παρά να πας να εργαστείς στο κατώτατο μισθό. Οπότε κάποιες γυναίκες ανειδίκευτες ή και ειδικευμένε με τον κατώτατο μισθό έχουν συμφέρον να μην εργάζονται γιατί έχουν ένα ελάχιστο εισόδημα, παίρνουν και οικογενειακά επιδόματα και συχνά στεγαστικά κλπ. Προστίθενται όλα αυτά τα επιδόματα και είναι σε καλύτερη μοίρα από ό,τι αν δούλευαν. Άρα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κοιτάξουν την κατάσταση αυτή των γυναικών αυτών και όπως σας είπα, δυστυχώς, στη δική μου χώρα έχουμε και τέτοιες καταστάσεις. Και έχουμε καταντήσει σε αυτό το σημείο που δεν υπάρχει περίπτωση να τις πείσει να εργαστούν αυτές τις γυναίκες. Αφήστε δε που αν έχουν και ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά ε, μικρής ηλικίας, πώς θα πάνε να εργαστούν αυτές οι γυναίκες. Τους βγαίνει και πιο φτηνά να κάθονται σπίτι και για την κοινωνία, να τους δίνουν ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα με οικογενειακά επιδόματα τέκνων, παρά αυτά τα δύο, τρία, τέσσερα παιδιά να πηγαίνουν και σε βρεφονιπιακούς σταθμούς για να δουλεύει η μαμά τους. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει, αν είναι σωστό. Να ε, βάζουμε τις γυναίκες σε μια τέτοια κατάσταση που να μην χρειάζεται καν να εργαστούν. Και όταν γεράσουν θα έχουν πάλι ένα ελάχιστο εισόδημα εγγυημένο που είναι περίπου το ε, αντίστοιχο με τον κατώτατο μισθό στη χώρα μου, 1.700 ευρώ. Στον κόσμο υπάρχει πλήθος ε, κόσμου που, που θα ονειρευόταν ένα τέτοιο μισθό. Και μας ενδιαφέρει αυτή η επιδοματική πολιτική ε, να μην μπορούν πια να απασχοληθούν αυτές οι γυναίκες τους κάνουμε χάρη, είναι υπηρεσία αυτή που τους προσφέρουμε. Άκουσα την κυρία Ματέρα να λέει ότι χρειάζονται λέει και ευρωπαϊκά επιδόματα και ενισχύσεις. Μεμονωμένα, τι εννοείται, δεν κατάλαβα. Ε, πώς μπορεί αυτό να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με 500 εκατομμύρια πολίτες πώς θα το οργανώσουμε αυτό. θα πρέπει όσο γενναιόδοροι και να είμαστε, να ξέρουμε, να μην ζητάμε τον ουρανό με mm. Μετά όμως νομίζω μάλλον ότι είναι προβλήματα μετάφραση. Δεν καταλαβαίνω την αιτιολογική σκέψη Β εγώ, όπου λέτε ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη οι ε, μόνοι γονείς στιγματίζονται και τα Τύπα, δίκτυα έχουν ένα ρόλο για την ενσωμάτωσή τους και θα πρέπει να αναγνωρίζονται. Τι θα πούν όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνω. Δεν βγάζει μεγάλο νόημα στα γαλλικά. Δεν ξέρω, ίσως το πρωτότυπο. Επίσης, στην αιτιολογική σκέψη Β, θα πρέπει να δώσουμε βάση στα διάφορα νομικά καθεστώτα. Γιατί μιλάμε για διάφορα επιδόματα. Μα αν παίρνουν επιδόματα, καλά κάνουν και τα παίρνουν. Μπράβο τους. Και αν είναι διαφορετικό το είδος από χώρα σε χώρα, ποιο είναι το πρόβλημα. Το σημαντικότερο δεν είναι ε, να είναι διαφορετικά τα επιδόματα, αλλά να παίρνουν. Το πρόβλημα θα ήταν να δεν υπήρχαν καθόλου. Να δούμε το νομικό καθεστώς στην αιτιολογική σκέψη Δέλτα. Είναι αυτό που λέει υποφελούνται από διάφορα είδη επιδομάτων. Ε, και ε, μήπως χρειάζεται λίγο να αναρμονίσουμε το οικογενειακό δίκαιο. Αυτό είναι άλλη ιστορία για τους μετανάστες ας πούμε. ή τις μετανάστριες. Επίσης, δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει ανήπαντρος γονέας ε, που δεν έχει εργασία αλλά είναι στο σπίτι, οικιακά. Τι είναι αυτό, άνεργοι γονείς που μπορεί να ζουν και σε ζευγάρι και δεν έχουν ε, επαγγελματική δραστηριότητα. Και κάποιος που μένει σπίτι του για να μεγαλώσει τα παιδιά του, αλλά έχει και σύντροφο. Τι εννοείται, δεν το έχω καταλάβει αυτό. και στην αιτιολογική σκέψη α, ε, ε, λατινικό. Ε, στα γαλλικά λέει ότι, στο θήτα μάλλον στο ελληνικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιέσεις διαδρομία είναι εντονότερες στις ηλικίες 25 έως 40. Τι θα πει αυτό. Μπορώ να καταλάβω τι εννοείται όταν είναι μικρά τα παιδιά κτλ. Αλλά πρέπει να ξαναδούμε τη γαλλική μετάφραση. Να την ξανακοιτάξουμε. Στη παράγραφο 5 τώρα ε, υπογραμμίζει την ανάγκη να διευκολυνθεί η πρόσβαση και τα λοιπά στην κατάρτιση. Οι οποίοι συχνά εγκαταλείπουν τις σπουδέ τους όταν μένουν έγκυες. Δεν θα πρέπει να πούμε αυτό. Θα πρέπει να λέμε να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να μην εγκαταλείπουν τις ε, σπουδές τους όταν μένουν έγκυες. Και να έχουν πρόσβαση στη μόρφωση, στην κατάρτιση, στην εκπαίδευση. Στο 8 γίνεται λόγος για κάποια επιδόματα ε, που τα χαρακτηρίζεται μάλιστα καθολικά. Τι θα ναι. πει αυτό καθολικά επιδόματα και για φορολογικές ελαφρύσεις και τα λοιπά ε, με βάση την εθνική νομοθεσία. Μάλλον λάθος τη μετάφραση είναι. Γενικά γνωρίζετε ότι οι ανήπαντρες μητέρες όταν είναι φτωχές ε, είναι στο φορολόγητο, δεν φορολογούνται. Οπότε τι φορολογικές ελαφρύνσεις από, από το μηδέν. Αυτό που ε, ε, στι γυναίκε τι οποίε θα μπορούσε αυτό να είναι χρήσιμο θα είναι σαν ύπαντρε μητέρε που έχουν μια λαμπρή σταδιοδρομία και μπορούν να αφαιρέσουν κάποια έξοδα γιατί εκπίπτουν ας πούμε τα έξοδα φύλαξη των παιδιών ή βρεφονιπιακή σταθμή, ακόμα και οικιακή βοηθός. Στη χώρα μου αυτό γίνεται. Άρα είχαμε ένα διευθυντή ε, στην εφορία που το είχε εισαγάγει αυτός ρύθμιση να μπορούν να υποφελούνται και οι άνδρες. Ήταν ο ίδιος ανήπαντρος και μάλλον τον συνέφερε. Αυτά τα ολίγα σχόλια είχα να κάνω και ε, νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να επανεξεταστεί η γαλλική μετάφραση. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε πολύ κυρία Λούλινγκ. Κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κυρία Ματέρα επέλεξε πολύ δύσκολο θέμα. <laughs> Όχι μόνο γιατί ο αριθμός των ανήπαντρων μητέρων αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, αλλά και γιατί για ολόκληρες δεκαετίες γίνονταν προσπάθειες να βρεθεί μια λύση για να βοηθηθούν αυτές οι γυναίκες και δεν πέτυχαν πολλές από αυτές. Όπως είπε και η κυρία Μπούρμαν, Πρέπει ίσως να λάβουμε υπόψη μας επίσης τους ανήπαντρους πατέρες που επίσης ασχολούνται με τα παιδιά τους, γιατί ο αριθμός των παιδιών που αναλαμβάνουν οι πατέρες μετά το διαζύγιο και αυτός αυξάνεται. Μερικοί από αυτούς τους πατέρες ε, αναλαμβάνουν τα παιδιά γιατί έχουν χειρεύσει. Μια άλλη δυσκολία είναι ότι οι επιπτώσεις αυτών των προβλημάτων τις υφίστανται τις επιπτώσεις τα παιδιά στην εκπαίδευση, στην ανατροφή τους γενικότερα. Αυτές οι γυναίκες ή αυτοί οι άντρες μπορεί να ζουν σε ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες ή μπορεί να την χάνει η οικογένεια ολόκληρη κοινωνικού αποκλεισμού και αυτό έχει δραματικές συνέπειες στη ζωή των παιδιών στη συνέχεια. Ίσως έχω επηρεαστεί από το γεγονός ότι είμαι και εγώ γιατρός. Αλλά όλα αυτά που είπε η κυρία Ματέρα αφορούν τις συνέπειες που έχει στη ζωή όλων η κατάσταση αυτή ανατροφής των παιδιών μόνον τους ή γιατί το κράτος δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του για να τους βοηθήσει. Εγώ ως ιατρός θα ήθελα στην έκθεση αυτή να μπει και το θέμα της πρόληψης ή για να μην φτάνουν σε αυτό το σημείο οι γυναίκες και οι άντρες. Το διαζύγιο συνήθως οφείλεται σε κάποιο κοινωνικό πρόβλημα όπως τον αλκοολισμό ή προβλήματα υγείας. Αν αυτά φανούν από νωρίς μπορεί να μην καταλήξουν μέχρι αυτές τις αρνητικές συνέπειες. Και κάτι ακόμα. Ε, Υπάρχουν πολύ γενναιόδορες προσφορές από την κοινωνία που πολλές φορές όμως την χάνουν χρήσεων Περιπτώσεις όπου μια γυναίκα δήλωσε ανήπαντρη μητέρα διότι έτσι την συνέφερε οικονομικά. Αν και είχε σύντροφο και συζούσαν αλλά επιλέγουν να μην παντρευτούν και δεν δηλώνουν καν ότι συζούν για να έχουν διπλά κοινωνικά ωφέλη. Μια τόσο γενναιόδορη πολιτική παρατηρείται όχι μόνο στη χώρα μου αλλά και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Πριν από 15 χρόνια το παρατήρησαν αυτό το φαινόμενο. και κατέληξαν ότι καλύτερα είναι η κοινωνία να στηρίζει τις οικογένειες πριν φτάσουν σε αυτό το σημείο και να ώστε να χρειάζεται τελικά να υποβοηθήσουν τις ανήπαντρες μητέρες. Και η κυρία Λούλινγκ ανέφερε ότι μερικές γυναίκες αποφασίζουν, επιλέγουν να μην παντρευτούν και να παραμείνουν ανήπαντρες μητέρες ίσως όμως να μην καταλαβαίνουν τι προβλήματα θα αντιμετωπίσουν. Επίσης στην Επιτροπή μας είπαμε ότι ο Σάτον Μάρτιο υπέβαλε μια έκθεση που μιλούσε για αυτά τα προβλήματα των γυναικών οι οποίες όμως δημιουργούν το 50% του πλούτου της κοινωνίας μας αλλά δεν ωφελούνται. γιατί δεν αναγνωρίζεται ούτε πληρώνεται καταλήλως η κατοίκον εργασία. Ή οι γυναίκες αναλαμβάνουν πολύ χαμηλοπληρωμένες δουλειές, κακοπληρωμένες, και δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Διότι αν τουλάχιστον οι γυναίκες αυτές πληρωνόνταν από την κοινωνία για την ανατροφή των παιδιών τους, Ίσως να τους αρκούσε αυτό για να μπορέσουν να πάρουν μία μερική τουλάχιστον εργασία, να κερδίσουν κάποια χαρήματα. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις και να γράψουμε και κάτι για την πρόληψη τέτοιων καταστάσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ζαμπόρσκα. Τώρα η Κομισιόν η κυρία Παρασκευά. Thank you, And, uh, thank you for... Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ ολόκληρη την Επιτροπή σας γιατί εξέτασε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που αν δεν απατώ με αφορά την ανέχεια και το κοινωνικό αποκλεισμό των γυναικών. Η Κομισιόν πάντως εδώ συμμερίζεται την άποψη ότι οι ανήπαντρες μητέρες δεν αποτελούν ομοιόμορφη κατηγορία κοινωνική. Από διαφορετικούς δρόμους φτάνουν σε αυτό το σημείο και υπάρχουν και διαφορετικές κατηγορίες ανυπάνδρων γυναικών. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα αν τι αντιμετωπίζουν οι ανυπανδρές μητέρες σε ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις γιατί έτσι η έκθεση θα συγκεκριμενοποιήσει την προσοχή της σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις. Τώρα, ως προς το τι ήδη λέει η έκθεση και όχι τι θα έπρεπε να προσθέσει, θα ήθελα να προσέξω ιδιαίτερα ορισμένες τροπολογίες, δηλαδή. Δυστυχώς ο αριθμός των ε, μονογονικών οικογενειών με βάση τα στοιχεία που έχουμε από το 2009 ε, έχει αυξηθεί κατά 48% έναντι 23% πριν από α, για τα ζεύγη με παιδιά. It should be highlighted uh, in the Commission's view in this report. Κατ' εμάς, το σημαντικότερο είναι πώς θα μπορούσαμε να συνδέσουμε την εξέβρεση μιας λύσης με τα υπάρχοντα προγράμματα πολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού όπως την Active Inclusion Strategy που προβλέπει επαρκή ελάχιστα εισοδήματα για να μπορούν όλοι να ζουν αξιοπρεπώς. Πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή σε οποιοδήποτε είδους δραστηριότητα υπάρχει away uh, from uh, labor market. Στην αγορά εργασίας και τρίτον και σημαντικότερον πρόσβαση σε ποιοτικές και οικονομικές enabling services που λέμε. Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για όλες τις οικογένειες, για τη στέγασή τους, για διάφορα. Και μια άλλη πολιτική που συνδέεται με αυτήν είναι εκείνη που αφορά την ανέχεια των παιδών. Το 2012 θα γράψουμε μία σύσταση πολέμησης της ανεχείας των παιδών και προώθησης της ευημερίας αυτών. Και σε αυτά τα πλαίσια θα στηρίξουμε τους γονείς που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ήδη η Ουγγρική Προεδρία έχει υποβάλει στο Συμβούλιο σχέδια συμπερασμάτων με στόχο να συγγραφεί αυτή η σύσταση ώστε οι, τα, οι μονογονικές οικογένειες να αντιμετωπιστούν. Η Κομισιόν συμφωνεί ότι το θέμα των μονογονικών οικογενειών είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά πρέπει να δούμε αν θα τονίσουμε ιδιαίτερα ή μόνο αυτούς που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις ή ολόκληρη αυτή την κατηγορία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ματέρα για να καταλήξει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακούστηκαν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα τις επόμενες μέρες είμαι βέβαιη ότι θα τα ξανασυζητήσουμε και σε ακόμα μεγαλύτερο βάθος. Θα υπάρχουν, θα κατατεθούν τροπολογίες, είμαι βέβαιη και θα έχουμε όλη την ευκαιρία να τις συζητήσουμε για να βελτιώσουμε την έκθεση. Προσπάθησα και σημείωσα μερικές από αυτές τις ιδέες και τις απαντήσεις και τα σχόλια που έκαναν οι συνάδελφοι, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα για να εξισορροπηθεί περισσότερο η έκθεση. Προσπάθησα, έκανα ό,τι μπορούσα. Δεν νομίζω ότι είναι παλαιομοδίτικη η έκθεση όπως είπαν μερικοί, γιατί εγώ προσωπικά συνομίλησα με όσο περισσότερες οργανώσεις μπορούσα και προσπάθησα να καταλάβω ακριβώς ποια είναι η κατάσταση των ανυπάνδρων γυναικών. Και από ό,τι είπαν οι συνάδελφοι αλλά και η Επιτροπή, καταλαβαίνω τώρα σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθώ. Πρέπει να σκεφτώ παραπάνω το θέμα της ε, ευάλω, του ευάλωτου του σημείου στο οποίο βρίσκονται αυτές οι ανήπανθερες γυναίκες γιατί θα τονίσω ακόμη περισσότερο από τη γενική κατηγορία την υποκατηγορία των ε, γυναικών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Θα θέλαμε βέβαια να γίνουν σούπερ γυναίκες και οι ενήπαντρες μητέρες, αλλά υπάρχει και το θέμα των πατέρων Ο τίτλος τελικά της έκθεσης αφορά μόνο τις ανήπανδρες γυναίκες. Δεν θα μιλήσουμε εδώ για τους άντρες. Αν χρειαστεί, τότε πρέπει να αλλάξουμε ολόκληρο τον τίτλο. Αν θέλετε να αλλάχθεί ο τίτλος για να συμπεριλάβουμε και τους ανήπανδρους πατέρες, με τα χαρά ε, το κάνω. Αλλά πάντως μιλούμε κυρίως για γυναίκες και μάλιστα ανήπαντρες μητέρες. Έχω μερικά στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι σχεδόν όλες οι μονογονικές οικογένειες αποτελούνται από γυναίκες. Υπάρχει και ένα ποσοστό ανυπάνδρων πατέρων, αλλά αν το συμπεριλάβω, το ξαναλέω, πρέπει να αλλάξω τον τίτλο της έκθεσης. Και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει οι πληροφορίες αυτές να δοθούν, να χορηγηθούν και στα κράτη-μέλη. Γιατί εδώ το θέμα είναι για το μέλλον όχι μόνο των γυναικών αυτών αλλά και των παιδιών τους και ιδιαίτερα η κυρία Ζαμπόρσκα είχε δίκιο. δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι πολλές από αυτές τις ανήπαντρες μητέρες είναι πολύ νεαρές ή έχουν υποστεί βία ή απλώς ε, τις εγκατέλειψε ο πατέρας των παιδιών τους και δεν έχουν άλλους πόρους. Πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη, να τα βοηθήσουμε να το καταλάβουν αυτό. Λυπάμαι που έφυγε η κυρία Λούλινγκ, γιατί ήθελα να της πω ότι εδώ δεν μιλάω για ευρωπαϊκά ταμεία. Μιλάω. Γιατί ξέρω ότι θα μου πει η Επιτροπή Προπολογισμών δεν έχουμε λεφτά. Εγώ μιλάω για ενθάρρυνση των χωρών μελών. Δεν λέω η Ένωση να χορηγήσει τίποτε πληρωμές τις ανήπαντρες μητέρες. Και ζήτησε αποσαφηνήσεις η κυρία Λούλινγκ γιατί είπα εγώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα άτυπο δίκτυο συνεννόησης των ανυπάντρων γυναικών. για να ενθαρρύνονται αυτές να επιστρέψουν στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Αυτό το λέω γιατί οι περισσότερες από αυτές είναι νεαρής ηλικίας και πελές από αυτές έχουν διακόψει τις σπουδέ των. Και επειδή είναι νεαρές θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν και μαθήματα πληροφορικής ή ξένων γλωσσών για να βελτιώσουν τα προσόντα τους γιατί αλλιώς είναι, δεν είναι ανταγωνιστικές στην αγορά εργασίας. Δεν είναι. Άλλος συνάδελφος, κύριε Γκουρμάη, είπε ότι πρέπει μερικά σημεία να τα εμβαθύνουμε περισσότερο, αλλά περιμένω να δω πρώτα ποιε είναι οι τροπολογίε των συναδέλφων για να δω τι να παραλείψω και τι να εμβαθύνω. Θα μπορούσα να είχα γράψει πολύ μακροσκελέστερη έκθεση αλλά δεν είχα το δικαίωμα γι' αυτό δεν τα είπα όλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ματέρα για την αλλαγή του τίτλου Νομίζω ότι δεν γίνεται. Λοιπόν, είναι έκθεση πρωτοβουλίας ε, που έτσι έγινε δεκτή. Αν μπορούσαμε να είχαμε αλλάξει την επικεφαλίδα και να την κάνουμε διαφορετική, για πανδρες μητέρες, τε και πατέρες, αυτό σημαίνει ότι δεν θα ήταν αρμοδιότητα της δικής μας Επιτροπής, αλλά της Επιτροπής Απασχόλησης και όχι ναι. της Επιτροπής Γυναικών. Οπότε πρέπει να το κρατήσουμε αυτό έτσι, χωρίς άνδρες. Ευχαριστώ για τη συζήτηση, πολύ ενδιαφέρουσα. Θυμίζω την προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών. 31 Μαΐου, 12 η ώρα το μεσημέρι, ακριβώς. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας κανονικά τον Ιούλιο, στη δε Ολομέλεια από Σεπτέμβρη. Έχουμε ένα τελευταίο σημείο στην ημερησία διάταξη, πριν περάσουμε στους συντονιστές, στις 7.30, ναι, που είναι άλλη συνεδρίαση, 17 και 30, στις 5.30. Και είναι ε, μια αναφορά της Αντιπροσωπείας Επιτροπής ε, Δικαιωμάτων και ισότητα των φίλων στην Βουδαπέστη. Ήταν η κυρία Γιαρόκα, η κυρία Κουρμάη και άλλοι συνάδελφοι και εγώ ίδια. Έχετε το πρόγραμμα ε, στους φακέλους σας, τι συζητήσαμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αυτού. Θα ήθελα να σας αναφέρω ορισμένα από τα θέματα που μας απασχόλησαν. Συναντηθήκαμε με τους αρμόδιους υπουργούς για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2011-2020. Μας μίλησαν για την οδηγία καταπολέμησης των διακρίσεων, ιδιαίτερα επέμεινε στα άτομα με αναπηρία. Επίσης, στήσαμε την οδηγία για τη μητρική άδεια, η άδεια μητρότητας και ο υπουργό μας είπε ότι δυσκολεύονται λίγο στο Συμβούλιο σε αυτό το θέμα. Και θα το διαβιβάσουν στην Πολωνική Προεδρία. Mm. Δεν θα τελειώσει επί Ουγγρικής Προεδρίας. Επίσης, συζητήσαμε και για τη στρατηγική 2020 ε, για τη βία, σεξουαλική βία για ε, το πρόγραμμα της Βακελόνης για τη φροντίδα των παιδιών και τη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη πολιτικών και οικονομικών από φάσεων. Μιλήσαμε και για το νέο ουγγρικό σύστημα. Είδαμε επίση και τους Υπουργούς Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ε, Θρησκευμάτων πολιτικών υποθέσεων και τα λοιπά που ασχολούνται και με την ισότητα των φύλων. Και για το νέο σύνταγμα πάλι συζητήσαμε εκεί και για τη στρατηγική ε, για τους Ρωμά. Συζητήσαμε για το mainstreaming στην πολιτική της Ουγγαρίας και το πρόβλημα της πορνείας και άλλα συναφή και σύμπαρο μαρτούντα. Αυτά συνοπτικά, θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι συναντήσαμε και έναν υφυπουργό ε, οικογενειακών υποθέσεων και την αρχή ε, ισότητας, κάποιου που είναι αρμόδιο για την ισότητα των αμοιβών και γενικότερα τα θέματα διακρίσεων. Και εκτός από όλους αυτούς συναντήσαμε και εκπροσώπους κοινωνίας των πολιτών και των πολιτριών. Είναι πολύ σημαντικό σε τέτοια ταξίδια αντιπροσωπείες να αφιερώνουμε πολύ χρόνο συναντήσεις με ΜΚΟ, κοινωνία των πολιτών, εκπροσώπους, ενώσεις, σωματεία και συλλόγους που μας περιγράφουν την κατάσταση στη χώρα τους επιτόπου. στα πλαίσια της Προεδρίας και τι περιμένουν, τι προσδοκίες και ελπίδες έχουν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τέλος, δώσαμε και συνέντευξη τύπου παρουσία πολλών δημοσιογράφων και δώσαμε και συνεντεύξεις ο καθένας έτσι μεμονωμένα, χωριστά. Δεν ξέρω αν θέλει να πάρει το λόγο κανένας άλλος συνάδελφος ή καμία που συμμετείχε. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα πριν περάσουμε στους συντονιστές. Όχι, δεν έχουμε. Ε, ωραία. Κυρίσω το πέρα συνεδρία της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συνεδρίαση, πολλές συζητήσεις και πολλές ή ψηφοφορίες. Λοιπόν, καλώς ορίζω τους συντονιστές. Περνάμε αμέσως στη συνεδρίαση των συντονιστών. Και όσοι δεν είναι συντονιστές, καλό σας βράδυ.